Ε, good Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας παρακαλώ, καθίστε. Θα ξεκινήσουμε σε ένα λεπτό. Έχουμε λοιπόν λίγο χρόνο για να καθίσουμε ο καθένας όσο πιο άνετα μπορεί και να ολοκληρώσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει. Ε, welcome. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους, κυρίως όμως την Επίτροπο και την υποδιορισμό και την ε, Αντιπρόεδρο για την Ενεργειακή Ένωση, την κυρία Αλένκα Μπρατούσεκ, η οποία είναι πρώην Πρωθυπουργός της Σλοβενίας. Η δημόσια αυτή ακρόαση έχει οργανωθεί από κοινού από τις Επιτροπές Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, τον συνάδελφο Τζοβάνι Λαβία Πρόεδρο και την και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Ήτρε, ε, ε, ε της οποίας εγώ είμαι ο πρόεδρος και βλέπετε εδώ μπροστά το όνομά μου, κύριος Μπούζεκ. Θα είμαστε και οι δύο συμπρόεδροι της ακρόασης αυτής. Επίσης θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στην αίθουσα αυτή, τα μέλη των δύο επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και εκπροσώπους των ευρωπαϊκών εταιριών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ε, από τα κράτη-μέλη, όπως επίσης πρέπει να πω ότι η δημόσια αυτή ακρόαση μεταδίδεται διαδικτυακά από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλοι λοιπόν οι Ευρωπαίοι που μας παρακολουθούν είναι και αυτοί ευπρόσδεκτοι. Θα ήθελα να πω ότι κάθε επιτροπή είναι εν γέννη υπεύθυνη για την ευρωπαϊκή πολιτική ενέργεια, την ασφάλεια της ε, προμήθειας ενέργειας, ε, την ε, εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την προώθηση της διασύνδεσης των ενεργειακών αγωγών και τη δημιουργία των διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των ε, υποδομών. Η ενεργειακή πολιτική θα είναι ένα σοβαρό θέμα στην ε, νομοθετική μας εργασία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για μας να ακούσουμε από την κυρία Αντιπρόεδρο, την υποδιορισμό επίτροπο, πώς σκοπεύει να χειριστεί τις δυσκολίες αυτές. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ζητήματα όπως ο ανταγωνισμός, οι εξωτερικές σχέσεις, ή τα θέματα της βιομηχανίας μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης. Όλοι σας, αγαπητοί συνάδελφοι, και από τις δύο επιτροπές και την ΕΝΒΙ και την Ήτρε έχετε πάρει, έχετε λάβει όλα τα έγγραφα. Το, την επιστολή ανάθεση στην κυρία ε, Επίτροπο, το βιογραφικό της σημείωμα, την δήλωση οικονομικών συμφερόντων και της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, όπως επίσης και τις γραπτές απαντήσεις στα ερωτήματά μας. υπάρχει το ερωτηματολόγιο με τις απαντήσεις στις θέσεις Και βεβαίως, πριν δώσω το λόγο στο συνάδελφο για να προεδρεύσει και αυτός, το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους υποδιορισμό επιτρόπους με βάση την, τις γενικές τους ικανότητες, την αφοσίωσή τους στην Ευρώπη και την προσωπική τους ανεξαρτησία. Επίσης, αξιολογεί τη γνώση του τομέα στον οποίο, τον οποίο θα αναλάβουν, όπως επίσης και τις δεξιότητές τους στον τομέα της επικοινωνίας. Ε, έχετε το λόγο κύριε συνάδελφοι. Ευχαριστώ κύριε Μπούζεκ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω την ε, υποδιορισμό επίτροπο και αντιπρόεδρο υπεύθυνη για την Ενεργειακή Ένωση, την κυρία Λένκα Μπράτουσεκ αφού διαδραμάτισε αρκετούς ρόλους ε, στο εσωτερικό της ε, ε, σλοβενικής κυβέρνησης, της σλοβενικής δημόσιας διοίκησης, ξεκίνησε την καριέρα της στο πολιτικό επίπεδο το 2011. Ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Σλοβενικού Κοινοβουλίου και το Φεβρουάριο του 2013 έγινε Πρωθυπουργός της Σλοβενίας. Πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός που ανέλαβε αυτά τα καθήκοντα. Το 2014 ανέλαβε και το Υπουργείο Υγείας. Ε, Στους τομείς της αρμοδιότητές της ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση του έργου διαφόρων επιτρόπων και κυρίως ε, του Επιτρόπου για την Κλιματική Αλλαγή και την Ενέργεια και του Επιτρέπου για το Περιβάλλον της θαλάσσιες πολιτικές και την αλία που καλύπτουν μεγάλο τμήμα των καθηκόντων του Επιτρόπου για το Περιβάλλον θα πρέπει να υπάρχει μια αποτελεσματική ενεργειακή ένωση με ε, σημαντικό ρόλο για την αλλαγή του κλίματος και θα πρέπει να καθοδηγήσει τις βασικές αρμοδιότητες και να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέτει και ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Θα είναι επίσης υπεύθυνη για την ανάπτυξη της ε, ε, θέσεων εργασίας της πράσινης ανάπτυξης και θέλει να κάνει την Ευρώπη ε, ηγέτη στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Γι' αυτό και ακριβώς και το χαρτοφυλάκιό της είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, στην οποία προεδρεύω. Εδώ και πολλά χρόνια δίνουμε μάχη για μια αποτελεσματική ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα και βιώσιμης ε, ε, ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ηγετικός ρόλος και πολύ καλά συντονισμένος Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες ε, παγκόσμιες διασκέψεις ε, για το κλίμα εν ώψη και της διάσκεψης των Παρισίων του 2015. Επίσης να υπάρχει και ε, κατάλληλη προοπτική για την ενέργεια και το κλίμα με ορίζοντα το 2030 και η ανάγκη φυσικά μεταρρύθμισης της αγοράς άνθρακα και το σύστημα ανταλλαγών εκπομπών, τα λεγόμενα ETS. Μετά από αυτά να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Μπούζεκ για να μας εξηγήσει λίγο πώς ακριβώς ε, θα γίνει η ακρόαση. Σας ευχαριστώ συνάδελφε, σας ευχαριστώ και για τα εισαγωγικά σας σχόλια και να σας πω το εξής. Στην αρχή της ακρόασης η υποψήφια επίτροπος θα κάνει μια εναρκτήρια δήλωση και Στην περίπτωση των ακροάσεων της Επιτροπής Ήτρε είχαμε 15 λεπτά για την ε, ομιλία, ενώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι 10 τα διαθέσιμα λεπτά. Συμφωνήσαμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στην υποψήφια Επίτροπο για 12 λεπτά. Ε, ένα ενδιάμεσο, ένα μέσος όρος μεταξύ των ε, δύο επιτροπών. Ενημερώθηκε η υποψήφια επίτροπος για την απόφασή μας, επομένως θα μιλήσει για 12 λεπτά. Αυτά στην αρχή. Στη συνέχεια, στο τέλος της ακρόασης θα της δοθούν 5 λεπτά για τις ε, καταληκτικές ε, ε, παρατηρήσεις της. Από εκεί και πέρα, ως συνήθως, θα έχουμε 45 λεπτά, 3 λεπτά για την κάθε ερώτηση, 1 λεπτό για την ερώτηση και 2 λεπτά για την απάντηση. Επίσης, να σας πω ότι για όλους τους συναδέλφους ισχύει αυτό και για την προτινόμενη επίτροπο, θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να σεβαστείτε το χρόνο αγόρευσης. Θα υπάρχουν 5 δευτερόλεπτα επιπλέον ανοχής για τους συναδέλφους και 10 δευτερόλεπτα για την υποψήφια επίτροπο και από εκεί και πέρα θα κλείνει το μικρόφωνο. Ορισμένε φορέ δεν είμαστε τόσο αγενεί, αλλά σε γενικέ γραμμέ έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Επομένω, είναι στο χέρι μας πριν ε, λήξει ο χρόνος, 10 δευτερόλεπτα πριν, θα αρχίσει να ανάβει ένα, ε, δύο αστεράκια στο τραπέζι. Επομένως, ε, κύρια προτινόμενη επίτροπε, θα δείτε ότι θα αναβοσβήνουν αυτά τα αστεράκια για να ξέρετε ότι ολοκληρώνεται ο χρόνος σας. Ο πρώτος γύρος ερωτήσεων θα είναι από εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Υπάρχει διερμηνία σε 23 γλώσσες, επομένως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μητρική σας γλώσσα. Σας παρακαλώ να μην μιλάτε πολύ γρήγορα, διότι πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διερμηνία. Η ε, συζήτηση μεταδίδεται ζωντανά από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορείτε να έχετε και πρόσβαση σε μαγνητοσκόπηση της ακρόασης ε, στην ίδια ιστοσελίδα. Ήγηκε η ώρα λοιπόν να ξεκινήσει η ακρόαση μετά από όλες αυτές τις αρχικές παρατηρήσεις ε, Κύρια Επίτροπε Υποδιορισμό, προ, τέος Πρωθυπουργέ, να σας δώσω το λόγο λοιπόν για να κάνετε τις αρχικές σας